Welcome, Καλώς ορίσατε αγαπητοί συνάδελφοι, καλώς ορίσατε στη σημερινή συνεδρία της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Πρωτού, καλώς ορίσουμε επίσημα τον Νίλ Στίγκεσεν, που είναι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Ας εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, αντιρρήσεις. Από ό,τι βλέπω δεν έχω να κάνω ανακοινώσει αλλά πρέπει να σας δώσω κάποιες πληροφορίες όσον αφορά τις τρέχουσες οργανικές διαπραγματεύσεις. Στις 25 Οκτωβρίου είχαμε τον δεύτερο τρίλογο για τον ΕΠΤΑ βάσει μια συμβαστική πρόταση από τον εισηγητή και τα τρία θεσμικά όργανα κατάφεραν να συμφωνήσουν για διάφορου ορισμού στα άρθρα 2, η Γενική Αρχή της Κατανομής στο άρθρο 18, παρακολούθηση των προϊόντων και διακυβέρνηση στο άρθρο 22, βιομετρική κίνδυνη στο άρθρο 42 και κυρώσει στα άρθρα 58 και 59. Μετά από περαιτέρω συζητήσεις δεν μπορέσαμε τουλάχιστον ακόμα να καταλήξουμε συμφωνία όσον αφορά την αδειοδότηση από την ΑΙΟΠΑ ή τις αρμόδιες εθνικές αρχές, συμπερίληψη των ΑΕΡΟΠΣ στις γενικές διατάξεις όσον αφορά την ελευθερία παροχής υπηρεσιών. Ο επόμενος πολιτικός τριμερής διάλογος προβλέπεται για τις 15 Νοεμβρίου. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον Ήλ Στιγκεσέν, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Όπως ξέρετε, το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δημιουργήθηκε μετά την έκθεση των πέντε προέδρων για την συμπλήρωση και την ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Βασικές αρμοδιότητες είναι αξιολόγηση της εφαρμογής του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αξιολόγηση της καταλληλότητας του δημοσιονομικού προσανατολισμού σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς επίσης και υποβολή προτάσεων για τη μελλοντική εξέλιξη του δημοσιονομικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τον Οκτώβριο το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο υπέβαλε τη δεύτερη της έκθεσή του. Η έκθεση αυτή αναθεωρεί τον τρόπο και εξολογεί μάλλον τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκε το δημοσιονομικό πλαίσιο για το 2017 και τονίζει θετικέ και αρνητικέ εξελίξει, καθώ επίση και τι δυνατότητε βελτίωση του πλαισίου αυτού. Προφανώ αυτά θα συζητήσουμε περαιτέρω και προτείνει όμω και η έκθεση αυτή και ε, Διάφορου τρόπου για την απλοποίηση του Συμφώνου σταθερότητα και ανάπτυξη και τη διακυβέρνησή του. Έρχεται λοιπόν την κατάλληλη στιγμή η έκθεση αυτή, καθότι συζητάμε και εμεί όλο και περισσότερο του δημοσιονομικού μα κανόνε, καθώ επίση και τι επιπτώσει τη μη συμμόρφωση με του κανόνε αυτού. Ξέρετε ότι σήμερα το Eurogroup θα συζητήσει τα εθνικά προσχέδια προπολογισμών και ξέρετε ότι έχουν προκύψει κάποια προβληματικά στοιχεία με ορισμένα κράτη-μέλη και τουλάχιστον με το κράτος αυτό το οποίο γνωρίζω καλύτερα. Έρχεται λοιπόν την κατάλληλη στιγμή η συζήτηση αυτή για τους δημοσιονομικού μας κανόνες. Θα ακούσουμε μια εισαγωγική παρέμβαση από τον καθηγητή Τίνγκεσεν και στη συνέχεια θα ακούσουμε τις ενδεχόμενες ερωτήσεις των μελών της Επιτροπής μας. Καλωσορίστε κύριε Τιγκεσέν, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σας αυτή. Στο Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο είχαμε και τη δυνατότητα πρώτερης ανταλλαγής απόψεων με τη δική σας την Επιτροπή και προσβλέπω και στην σημερινή μας ανταλλαγή απόψεων. Υπενθυμίσατε κύριε Πρόεδρε στα μέλη μας ποια είναι η εντολή μας. Βρισκόμαστε στην θέση εκείνη την εύκολη ουσιαστικά θα έλεγα όπου καλούμεθα να συζητήσουμε τα έχω συμβεί στο παρελθόν και συγκεκριμένα στο έτος 2017 και από την άλλη όμως μπορούμε να κάνουμε και προτάσεις για το πώς θα πρέπει να εξελιχθούν τα πράγματα στο μέλλον, ιδίως πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τους κανόνες οποίους έχουμε. Επομένως μπορούμε εκ των υστέρων εμείς να κάνουμε κάποιες προτάσεις για τόσο έχουν συμβεί ή έχουμε ακόμα και τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιες πιο ελεύθερες, αν θέλετε, προβλέψεις και εκτιμήσεις για τις μελλοντικέ εξελίξεις, πώς μπορούμε δηλαδή να ολοκληρώσουμε και να βαθύνουμε καλύτερα την Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Επομένως, αν είμαστε πολύ επικριτικοί ορισμένες φορές ή αν κάνουμε, αν θέλετε, α, πολλές προτάσεις για το μέλλον, αυτό είναι άλλωστε και ο ρόλος μας. Στην έκθεση αυτή κάνουμε μια λεπτομερή αξιολόγηση του 2017, αφού το ανέφερα πριν από λίγο. Θεωρούμε ότι το έτος αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι το πρώτο έτος κατά τη διάρκεια του οποίου είχαμε μια σημαντική πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη μετά την κρίση η οποία είχε, εντάθηκε κυρίως το 2012-2013, όπου είδαμε μια πολύ έντονη ύφεση. Προτού επισέλθουμε σε περισσότερες λεπτομέρειες και προτού κάνουμε κάποιες επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόστηκαν οι κανόνε του 2017, θα ήθελα να σα πεθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ουσιαστικά υποστηρίζει το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωση. Χρειαζόμαστε το πλαίσιο αυτό, χρειαζόμαστε του κανόνε αυτού προκειμένου να μπορούμε να έχουμε στα πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης συγκεκριμένους κανόνες και να μπορούμε να διορθώνουμε σφάλματα που γίνονται στη δημοσιονομική πολιτική και να αποφεύγουμε τελικά ακόμα και αποκλήσεις ή δευτερογενείς συνέπειες της μη συμμόρφωσης με τους κανόνες αυτούς. Σε ένα μεγάλο βαθμό έχουμε επιτύχει το στόχο αυτό μετά την οικονομική κρίση. Ήδη στην προηγούμενη ετήσια έκθεσή μας για το 2016 ήμασταν πιο θετικοί στα σχόλιά μας. Είμαστε λιγότερο θετικοί για το 2017 και αυτό διότι οι οικονομικές προοπτικές ήταν πιο θετικές για το 2017. Επομένως θα μπορούσαμε να τα είχαμε πάει και ακόμα καλύτερα. Και από ό,τι φαίνεται οι προοπτικές αυτές συνεχίζονται και για το 2018 και ελπίζω και για το 2019. Και όπως συζητήσαμε ήδη και στην έκθεση του Ιουνίου, ο δημοσιονομικός προσανατολισμός για το 2019 φαίνεται να είναι θετικός. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το 2017 έδωσε μία περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία και αυτό δίκησε βέβαια σε κάποιες τάσεις ενισχυτικές των κυκλικών τάσεων. Και δυστυχώς αυτό το είδαμε κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν υψηλό δημόσιο χρέος. Το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο δεν θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρχει αναγκαστικά μια πολύ αυστηρή εφαρμογή των κανόνων. Αναγνωρίζουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κάποια διακριτική ευχαίρεια για τα κράτη-μέλη, αλλά αυτή η διακριτική ευχαίρεια και ευελιξία ήταν ε, ιδιαίτερα, αν θέλετε, υπερβολική το 2017. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε κάποιες σχετικές συστάσεις. Ξέρουμε ότι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει από κοινού την ευθύνη για την εφαρμογή των κανόνων με το Συμβούλιο και είχε και την υποστήριξη του Συμβουλίου στις συστάσεις της. Βέβαια, το Συμβούλιο σε περαιτέρω συστάσεις που έκανε μετά τις προτάσεις Ευρωπαϊκή Επιτροπής επανήλθε σε κάποιε από τι προτάσει που έκανε αρχικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε πιο επικριτικοί και να προωθήσουμε μια γενικότερη αναθεώρηση των κανόνων προκειμένου να περνούμε σε επιμέρους κάθε φορά διορθώσεις και προσαρμογές για κάθε χώρα ξεχωριστά σε ένα σύστημα το οποίο είναι ήδη πολύ πολύπλοκο. Ας δούμε τώρα τι λέμε στα κεφάλαια 2, 3 και 4, αναφερόμαστε εδώ πέρα στο 2017. Πέρα από τα όσα σας είπα, προσπαθούμε εδώ πέρα να αναφερθούμε και στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και βλέπουμε επίση και ποιε είναι οι συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά το δημοσιονομικό προσανατολισμό του 2017. Στα δύο τελευταία κεφάλαια ατενίζουμε, αν θέλετε, περισσότερο στο μέλλον. Προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η γενικότερη εμπειρία που έχουμε ήδη από το 2015 με το καθεστώς ευελιξίας και στο κεφάλαιο 6 αναφερόμαστε στην μελλοντική εξέλιξη του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου και του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Α δούμε τώρα ποιε είναι οι βασικέ συστάσει που γίνονται στην έκθεση αυτή. Η πρώτη σύσταση που γίνεται είναι ότι καταρχάς έχει πρώτη διαπίστωση μάλλον ότι έχει βελτιωθεί η οικονομική κατάσταση στην Ευρωζώνη το 2017 σε σχέση με τα παρελθόντα έτη. Βλέπουμε επίσης ότι το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης δεν προσαρμόστηκε στις καλύτερες οικονομικές συνθήκες και αυτό γιατί υπήρχε μια ασυμμετρία όσον αφορά τους κανόνες και δεν προβλεπόταν ε, η απαραίτητη διόρθωση κάθε φορά που οι συνθήκες βελτιώνονταν. Και βλέπουμε επίσης ότι η διακριτική ευχέρεια που χρησιμοποιήθηκε για το μετριασμό των απαιτήσεων ουσιαστικά δεν βοήθησε την γενικότερη συμμόρφωση με τους κανόνες. Και βλέπουμε ότι για αυτό το λόγο οδηγηθήκαμε ουσιαστικά σε κάποιες καταστάσεις όπου τα κράτη-μέλη απέκλαν τελικά από τους κανόνες. Επίσης είχαμε μία ανάποδη χρήση των εκτάκτων, αν θέλετε, προσδόκητων εσόδων που προέκυψαν κατά το 2017. Τα έσοδα αυτά δεν χρησιμοποιήθηκαν με εναρμονισμένο τρόπο και οι χώρες οι οποίες τελικά είχαν θετικά οικονομικά αποτελέσματα αποφελήθηκαν και κατάφεραν ουσιαστικά να εξηγιάνουν περισσότερο τα δημόσια οικονομικά τους, ενώ χώρες εκείνες οι οποίες είχαν υψηλότερο χρέος τελικά δαπάνησαν τις τα αυτά έσοδα χωρίς να τα χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν την οικονομική τους κατάσταση. Συναλλικά μπορούμε να πούμε ότι υπήρχε κατάλληλη δημοσιονομική εξυγίανση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο κρατών μελών, σε εθνικό επίπεδο, Υπήρχαν πολλέ χώρες οι οποίες τελικά δεν εκμεταλλεύτηκαν σωστά την ευκαιρία που τους δόθηκε προκειμένου να βελτιώσουν την κατάσταση του χρέους τους και να δημιουργήσουν τα απαραίτητα δημοσιονομικά αποθέματα. Το Νοέμβριο του 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μία δημοσιονομική καθοδήγηση και πρότεινε τότε να υπάρχει μια επιπλέον δημοσιονομική επέκταση της τάξης του 0,5% όσον αφορά το συλλογικό ΑΕΠ. Εμείς θεωρήσαμε ότι δεν ήταν δικαιολογημένο κάτι τέτοιο ούτε εκείνη την εποχή, μολονότι οι πληροφορίες οι οποίες είχαμε τότε δεν ήταν ολοκληρωμένες, αλλά ούτε εκ των υστέρων ήταν δικαιολογημένη μια τέτοια σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθότι τελικά δεν συμμορφωνόταν με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Επίσης, ε, η σύσταση αυτή έστειλε κάποια παραπληντικά μηνύματα προ τα κράτη-μέλη τη στιγμή εκείνη που θα έπρεπε ουσιαστικά να ασχολείται περισσότερο με την ενίσχυση τη δημοσιονομική εξυγίανση. Και ουσιαστικά οι ρήτρε ευελιξία που χρησιμοποιήθηκαν το 2017 θα έχουν εφαρμογή τελικά μόνο για το 2018. Επίσης, τα ανεξάρτητα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια πετύχαν τις περισσότερες φορές να ενισχύσουν την όλη συζήτηση για τα δημόσια οικονομικά και να ενισχύσουν την δημοσιονομική εποπτεία. Αυτό έγινε στη Ρουμανία για παράδειγμα και την Ιταλία όπου τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια της χώρας των χωρών αυτών επέκριναν τις δημοσιονομικές προοπτικές που επίσημα υπέβαλαν οι χώρες αυτές. Τα δημοσιονομικά αυτά συμβούλια στις υπόλοιπες χώρες όμως δεν τοποθετήθηκαν, ίσως επειδή έχουν και τελικά περιορισμένους πόρους, δεν έχουν την απαραίτητη πρόσβαση σε πληροφορίες και τέλος επειδή τα Ινστιτούτα αυτά δεν συμμετείχαν σε συζητήσει εκείνε που γίνανε μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, κρατών μελών. Επομένω, ε, ακόμα και αν είχαν να κάνουν κάποιε συστάσει, τελικά αυτέ δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στην επίσημη συζήτηση που γίνεται μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κρατών μελών. Μία ακόμα σύσταση που γίνεται στην έκθεση έχει να κάνει με την απλούστευση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη. Λέμε ότι έχουν γίνει απόπειρε προκειμένου το σύμφωνο αυτό να γίνει πιο ευέλικτο και πιο αποτελεσματικό. Αλλά δυστυχώ οι απόπειρε αυτέ δεν έχουν ε, εφαρμοστεί από όλα τα κράτη-μέλη με τρόπο συστηματικό. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνει μια γενικότερη αναθεώρηση του Συμφώνου Σταθερότητα και Ανάπτυξη και επίση του συστήματο διακυβέρνησή του. Στην τελευταία αυτή διαφάνεια, στη σελίδα 6 τη παρουσίασή μου, βλέπετε ότι προτείνουμε ουσιαστικά να επιστρέψουμε σε έναν βασικό στόχο των δημοσιονομικών κανόνων που να έχει να κάνει με τη μείωση του δημοσίου χρέους και να χρησιμοποιείται ένα βασικό μέσο για να το πετύχουμε αυτό, βασικά να είναι ο δείκτης για τις δημόσιες δαπάνες. Να γνωρίζουμε δηλαδή ποιες είναι οι καθαρές δημόσιες δαπάνες, αν υπάρχει αύξησή τους και αν η αύξηση αυτή τελικά συμμορφώνεται με τους γενικότερους δημοσιονομικούς στόχους για τη χώρα αυτή και με τη γενικότερη οικονομική ανάπτυξη θεωρούμε ότι υπάρχουν ε, αρκετοί οι οποίοι υποστηρίζουν την προσέγγιση αυτή. Ήδη από το 2016 ανάλογο έχει πει, μια ανάλογη πρόταση έχει κάνει και η Ολλανδική κυβέρνηση, αλλά και οργανισμοί όπως ο ΩΣΑ ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εμείς κάνουμε εδώ μια πιο συγκεκριμένη πρόταση και λέμε ότι ένα τέτοιο σύστημα βέβαια απαιτεί ένα βαθμό ευελιξία σε βάθος χρόνου, δεν μπορεί να εφαρμόζεται κατά αυτόν τον τρόπο σε κάθε αλλά προτιμούμε από το να έχουμε έναν μονοετή οικονομικό κύκλο να μπορούμε να θα περισσότερο σε έναν τριετή οικονομικό κύκλο. Και λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διακριτική, αν θέλετε, μια εντελώ ξεχωριστή στάση απέναντι στην οικονομική ανάλυση μια χώρα και των πολιτικών αποφάσεων που μπορούν να λαμβάνονται για μια χώρα. Και ότι θα πρέπει αυτό να είναι πάντα σαφέ. Σα ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ολοκληρώνω εδώ την παρουσίασή μου. Βλέπετε ότι υπάρχουν και άλλοι πίνακε και άλλε διαφάνειε, τι οποίε δεν σα έχω παρουσιάσει. Σα δίνουν τη δυνατότητα να επισέλθετε σε περισσότερε λεπτομέρειε, σε μια πολυσύλλευη τελικά έκθεση. Και νομίζω ότι αυτό θα μπορούσε να εμπλουτίσει και τι συζητήσει που θα κάνετε εσεί εδώ στην Επιτροπή σα. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ήταν ξεκάθαρος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα με τους συναδέλφους βουλευτές. Πρώτη εκ μέρους του ΕΛ και Ντανόντα Χούπνερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Καθηγητά, θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα της διακυβέρνησης που αναφέρατε στο τέλος ε, της παρέμβασής σας, ε, διότι βλέπετε τους δύο ρόλους ε, τους οποίους αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τους μεσονομικούς κανόνες θέλετε να τη δείτε ως έναν μέρο του θεματοφύλακα αλλά και ως εκτελεστική εξουσία, άρα έχει και πολιτικό ρόλο η Κομισιόν ε, καθότι εξολογεί τα δημοσιονομικά σχέδια και διατυπώνει συστάσεις. Στην έκθεση υπάρχει δυνητική σύγκρουση συμφερόντων στο πλαίσιο αυτό. Έχω το εξής ερώτημα. Όταν ε, αναφέρατε δύο δυνατότητες, είπατε ότι στο πλαίσιο Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα ξεχωριστό, μια ξεχωριστή λειτουργία, ε, ανεξάρτητη, αυτή είναι μια επιλογή, σαν ένας κλειστός χώρος, ενώ η δεύτερη δυνατότητα θα ήταν μια εξωτερική ανάθεση οικονομικών αναλύσεων σε έναν περισσότερους εξωτερικούς ε, φορείς. Αλλά δεν κάνετε κάποια πρόταση, δηλαδή ποια από τις δύο επιλογές θα προτιμούσατε και δεν ξέρω και αν έχετε κάποια προσωπική άποψη. Πόσα λεπτά έχω, πέντε, λίγο πολύ. Έχεις και 30 δευτερόλεπτα για ένα συμπληρωματικό ερώτημα, για να μπορείς να απαντήσει Ναι, αυτή η αλλαγή του κανόνα ε, evidence-based, μετά λέτε για μια οροφή που πρέπει να είναι κάτω από αυτή είναι οι δημόσιες δαπάνες, προβλέπετε διεξαιρέσεις, μιλάτε μεταξύ άλλων για οικονομική ύφεση. Πώς όμως τη βλέπετε την εξαίρεση αυτή σε σχέση με τις οικονομικές, ε, οικονομική ύφεση. Δηλαδή πώς μπορούμε να προστατεύσουμε σε μια τέτοια περίοδο ύφεση ε, και με το σύστημα που προτείνεται στις στρατηγικές επενδύσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις δυο σας αυτές ερωτήσεις. Ναι, πράγματι δεν εξέφρασα ρητός μια προτίμηση, γιατί υπάρχουν επιχειρήματα που στηρίζουν και την μεν και την δε. Αυτό ο η κλειστή ανάθεση του αναλυτικού έργου σε μια ξεχωριστή αρχή, ίσως στο πλαίσιο της Κομισιόν, είναι κάτι ριζοσπαστικό. Σίγουρα μπορεί να ασκεί ε, επιτήρηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και άλλοι διεθνείς φορείς θα μπορούσαν να το κάνουν. Το βλέπουμε στο εξωτερικό, ίσως όχι τόσο ξεκάθαρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βέβαια έχουμε και τη συμμόρφωση με την χρήση των πόρων και τη τύπωση συστάσεων εκ μέρους της Κομισιόν. Η άλλοι είναι κάπως πιο συζητήσιμη. Πρώτα στα αναφέρουμε όμως γιατί συζητείτε Και επισήμως από ό,τι φαίνεται, αλλά κάποια έτοιμη λύση δεν βλέπουμε. Άρα η προσωπική μου άποψη, αν αυτό με ρωτάτε, είναι ότι η πρώτη επιλογή είναι πιο ρεαλιστική, η δεύτερη είναι μια επιλογή η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της όλης συζήτησης που έχει ξεκινήσει και θα μπορούσε και αυτή να ληφθεί υπόψη. Σε ό,τι αφορά αυτό το κριτήριο αναφοράς για τις δημόσιες δαπάνες, είναι πράγματι αφορά το σύνολο των δαπανών, δεν γίνεται διάκριση μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών δαπανών. Σε ό,τι αφορά τους μοσομικού κανόνες, το μεγαλύτερο μέρος τους βλέπουμε αδοποιημένα τις δαπάνες. Βέβαια σήμερα ήδη γίνονται απόπειρε προστασίας μετά τις περικοπές που είδαμε το 2013 και μετά δεν απέδωσαν όλα αυτά τα μέτρα και τόσο καλά. Άρα το 2017 που αναλύσαμε δύο χώρες είδαμε ότι χρησιμοποίησαν ε, αυτό το ειδικό ε, επίδομα για τις επενδύσεις επειδή υπήρχε αυτή η δυνατότητα αυστηρό σύστημα ίσως δεν, το πιο αυστηρό σύστημα να μην λειτουργεί τόσο καλά. Εμείς στην ε, έκθεσή μας περιοριστήκαμε πιο πολύ στα ομαδοποιημένα μεγέθη, αλλά σίγουρα θα πρέπει οι επενδύσεις να προστατευτούν καλύτερα στο μέλλον από ό,τι στη διάρκεια της κρίσης. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρέσου. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις αυτές που μας δώσατε. η δημοσιονομική ανάλυση θα πρέπει να είναι καλύτερη από την πολιτική ανάλυση, σας λένε. Παράλληλα, το δημοσιονομικό έτος το 2017 ήταν καλύτερο και αν ήταν καλύτερο θα είχαμε ε, αποτρέψει τα αποτελέσματα, τα εκλογικά που είδαμε στην Ιταλία. Νομίζω ότι σε όλα αυτά χρειάζεται και κάποια προσοχή για τη συνέχεια του δημοσιονομικού συμφώνου. Νομίζω ότι ξεκινάει μια συζήτηση η οποία είναι πλήρη εξελίξη και νομίζω ότι όλοι αναγνωρίζουμε ότι κάτι θα πρέπει να γίνει. Κάτι θα πρέπει να γίνει για να αναδιαμορφωθεί η διάταξη αυτή, η ομάδα αυτή διατάξεων. Ένα κώδικα ε, σύγκληση είναι αυτό που σκεφτόμαστε και γιατί αυτό που μα απασχολεί βασικά είναι ότι θα πρέπει να επιτρέπουμε στα κράτη να προγραμματίζουν τη δημοσιονομική τους στρατηγική σε ένα πιο μακροπρόθεσμο επίπεδο και όχι μόνο αναδημοσιονομικό έτος. Αυτό ως ιδέα θεωρείτε ότι συγκαταλέγεται στις αρχές ε, επί των οποίων θα μπορούσατε να εργαστείτε. Ένα δεύτερο στοιχείο το οποίο θα ήθελα να θέσω. Μία σκέψη, μία ανησυχία. Κυρία Χούμπνερ, είπατε ότι σας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Ε, εμένα αυτό που με απασχολεί ιδιαίτερα πέρα από τον κανόνα είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την βιώσιμη ανάπτυξη πιο συγκεκριμένα. Αυτό με απασχολεί ιδιαίτερος και κατά πάσα πιθανότητα δεν λήφθη επαρκώς υπόψη στην ε, κατάρτιση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά και την δημοσιονομική ικανότητα τη Ευρωζώνης, πιστεύετε πώς πιστεύετε ότι θα πρέπει να διαμορφωθεί στο μέλλον η διαχείριση και η διακυβέρνηση τη Ευρωζώνης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μπερές. Θεωρούμε ότι η εντολή μας επικεντρώνεται στην ε, μεταρρύθμιση του Συμφώνου σταθερότητα ε, και Ανάπτυξης. Αυτή είναι, αυτός είναι ο σκοπός και η πρόθεση. Και αν κοιτάξετε την εντολή μας πώς διαμορφώνεται, δεν έχουμε εξετάσει το πιο θεμελιώδης ζήτημα του κώδικα σύγκλησης, το οποίο περιλαμβάνεται, το οποίο αναφέρεται μάλλον. Κανείς δεν αμφιβάλλει φυσικά για τη σημασία αυτού. Αλλά υπάρχει μια διάκριση στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ των δημοσιονομικών κανόνων, όπου υπάρχει αξιολόγηση και θέλουμε να κοιτάξουμε προκειμένου να μην προκληθεί περαιτέρω απόκληση και το θέμα της γενικότερης σύγκλησης και αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ε, ατζέντα. Όχι τόσο όμως τμήμα της δικής μας ατζέντα, ε, αν και το αναφέρουμε στην ε, έκθεσή μας. Για τι επενδύσει και τον προγραμματισμό των επενδύσεων. Είναι Πολύ σημαντικό θέμα αυτό. Και αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να δοθεί ένα περιθώριο λιγμού στα κράτη-μέλη για τι επενδύσει του και για τι προτάσει συντηρητικών μεταρρυθμίσεων κτλ. Υπάρχουν δύο δυνατότητε και δεν υπήρχε ποτέ ιδιαίτερη υποστήριξη για ένα χρυσό κανόνα προστασία των επενδύσεων γιατί αυτό περιλαμβάνει πολλά και γενικά πράγματα. Τελευταία επικεντρωνόμαστε στην ε, οικοδόμηση συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω του προγράμματος ε, Juncker. για να ξεπεράσουμε τα αυστηρά δημοσιονομικά μέσα. Αυτό θα Μα έβρισκε σύμφωνους. Δεν το έχουμε συζητήσει όμω και δεν είμαστε και ειδικοί για το θέμα αυτό. Σε ό,τι αφορά την επιβολή τέτοιων σχεδίων ε, επενδύσεων. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει εσεί να απαντήσετε την τρίτη ερώτηση. Ο πρόεδρο. Ευχαριστώ. Θέλετε να κάνετε επερώτηση, η κυρία Περές. Ναι, για την δημοσιονομική ικανότητα, παρακαλώ. Όπως αναφέραμε και στην έκθεσή μας πέρσι το καλοκαίρι, το καλοκαίρι μάλλον, μας αρέσει αυτή η ιδέα για τη δημοσιονομική ικανότητα. Νομίζω ότι αν ένα πράγμα μας έχει διδάξει η κρίση, είναι ότι υπάρχουν καταστάσεις όπου ακόμα και οι πιο αυστηροί δημοσιονομικοί και νομισματικοί πολιτικοί δεν μπορούν να εξασφαλίσουν μια σταθερή ανάπτυξη. Είμαστε λοιπόν από τις αρχές υπέρ μια κεντρική δημοσιονομική διαχείριση. Αλλά κατανοούμε ότι για να εγκριθεί αυτό και να περάσει αυτό πολιτικά θα πρέπει να λειτουργούν και οι εθνικοί κανόνε. Και εδώ υπάρχει μία αναλογία με την συζήτηση που γίνεται για την Τραπεζική Ένωση και για την κατανομή του κινδύνου, την καταμερισμό του κινδύνου. Θα πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι αυτά τα δύο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτή η κεντρική δημοσιονομική ικανότητα θα πρέπει να ακολουθεί την προϋπόθεση του να τηρούνται οι εθνικοί δημοσιονομικοί κανόνες. Προκειμένου λοιπόν να μην υπονομεύεται η προθυμία των κρατών να ακολουθούν τέτοιου κανόνες, θα πρέπει να δοθούν πιο πολύ κίνητρα. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα σταθεροποίηση επενδύσεων είναι πολύ περιορισμένη σε ό,τι αφορά την προοικοδότησή τη. Θα πρέπει να αυξηθεί το σχετικό κονδύλι και ανησυχούμε γιατί θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναβάλει τη συζήτηση αυτή και η συζήτηση αυτή θα ξεπεράσει τα όρια του επόμενου έτους. Υπάρχει λοιπόν μια άλλη λεξάρτηση μεταξύ κεντρικής οικονομικής ικανότητας και των κανόνων. Ο κύριος Λούκες, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας, θα μιλήσω γερμανικά. Καλώς ορίσω καταρχάς. Καλώς ορίσω καταρχάς την πρώτη σας για να υπάρχουν ανεξάρτητες επιτροπές για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εξαιρέσεων και παρεκκλήσεων. Αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό αλλά κοιτάω και τους νέους ε, δημοσιονομικούς ε, κανόνες σας. Πιστεύω ότι είναι υπερβολικά χαλαρά τα πράγματα. Είναι προβληματικό, πιστεύω, να υπάρχει ένα τριετές πρόγραμμα εποπτείας, γιατί κανονικά μετά από τα πρώτα τρία χρόνια θα πρέπει να υπάρχει μόνο μία προειδοποίηση και μετά από έξι χρόνια να υπάρχει α, δυνατότητα κυρώσεων. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ χαλαρό. Γιατί δείχνετε τέτοια γενναιοδορία, εξηγήστε μα. Είμαι πολύ επικριτικός επίση, σε ό,τι αφορά την πρότασή σα για τον δημοσιονομική α, δικλείδα για το θέμα του χρέους του 60% γιατί έχουμε και το κριτήριο του 3% για το έλλειμμα. Αυτό τι το κάνετε, το α, καταργείται. Δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή κυριώσεων και οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες δεν προβλέπουν κυρώσεις. Δεν φαίνεται είναι αυτό στην ε, έκτασή σας. Άρα τι κανόνες εφαρμογής έχετε υπόψη σας. Θέλετε να υπάρχει δυνατότητα να επιβάλλονται κυρώσεις ή τις καταργείτε και αυτές. Με την πρότασή σας, επόμενη ερώτηση. Πείτε μου παρακαλώ για την πολιτική δαπανών. Εδώ βάζεται ως κριτήριο το, την ανάπτυξη των δαπανών και την αυτόματη λειτουργία σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι βασικά είναι αυτόματη δαπάνη κονδυλίων. Τα χρήματα όμως αυτά δεν θα πρέπει να δαπανώνται με παραγωγικό τρόπο. Πώς μπορούμε λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η μονομερής ε, παροχή κινήτρων θα προωθήσει ε, εύλογα παραγωγικά έργα για την μακροοικονομική ανάπτυξη που χρειάζεται σε περίπτωση κρίσεων. Χρειάζεται λοιπόν εγγύηση για την ποιότητα των επενδύσεων και θα καλωσόριζα λοιπόν ενδεχομένως κάποιο κανόνα σχετικά με αυτό. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας κύριε Λούκε και έχετε δίκιο ότι θέλουμε να δώσουμε ε, παρόλα αυτά έμφαση ιδίως στο δομικό έλλειμμα uh, Υπάρχει αυτό το 3%. Στόχος έχει να υπάρχει κάποια αξιοπιστία. Είναι κάτι που το γνωρίζει ο κόσμος. Αλλά μπορεί να θεωρείται και κάπως αυθαίρετο ή ένας εύκολος στόχος, όπως βλέπουμε στο σημερινό περιβάλλον. Το 3% εύκολα το έχουν επιτύχει σχεδόν όλες οι χώρες, παρά την επισφαλή συχνά κατάσταση των δημοσίων οικονομικών ορισμένων εξ αυτών. Άρα εστιάζουμε στη μείωση του χρέους, έχουμε το 6% ως, το 60% όριο και δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι θα είναι εύκολο, ότι μπορεί να επιτευχθεί αυτό μέσα σε 15-20 χρόνια, αλλά αυτή είναι η που πρέπει να ακολουθήσουμε. Αυτό το ρυθμό προσπαθούμε να αναπτύξουμε με το τελευταίο κεφάλαιο. Δεν είναι και πολύ ήπιο μέτρο, ίσως πιο ήπιο βέβαια είναι για κάποιες χώρες γιατί επιτρέπει ε, πιο αυτόματη σταθεροποίηση από ότι οι υφιστάμενοι κανόνες και στο τελευταίο κεφάλαιο κάνουμε και κάποιες συγκρίσεις για τη μετάβαση που δεν ήταν τόσο απότομη. Είναι όμως μια εκδοχή που δεν είναι και τόσο ήπια γιατί θα απαιτήσει θετικά δημόσια πλεονάσματα για κάποια χρόνια στις χώρες που είναι ιδιαίτερα χρεωμένες. Σε ό,τι αφορά το net expenditure growth, είναι ένα ομαδοποιημένο σε ένας ομαδοποιημένος δείκτης δεν κάνει κάποια διαφοροποίηση ούτε περιορίζει κάπου στα κράτη-μέλη ε, σε ό,τι αφορά το πού θα δαπανίσουν ε, αν θέλουν να επιβάλλουν περισσότερους φως μπορούν να το κάνουν. Αλλά αν υπάρχει μεγάλη μείωση της φορολόγησης θα πρέπει να υπάρχει μείωση και των δαπανών. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η δημοσιονομική απέτηση θα έχει κάποιες επιπτώσεις και σε ό,τι αφορά τον κάνω του 3%. Θα είναι ίσως πιο αποδεκτό με τρόπο πολιτικής πλευράς. Εσείς θα κρίνετε καλύτερα βέβαια. Και βέβαια μπορούμε να λάβουμε υπόψη μας και κάποιες παραμέτρους ποιότητας εδώ. Επιτήρηση λοιπά. Δύσκολο όμως αυτό μπορεί να περιληφθεί στους κανόνες. Αυτή ως απάντηση. Μα δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου για τις κυρώσεις, κύριο Λούκε. Ουσιαστικά τις καταργεί την de facto, γιατί δεν υπάρχει μηχανισμός ένισης. Τι είπατε? Α, ότι καταργούμε τις κυρώσεις. Όχι, τη συσχετίζουμε με αυτό το νέο σύστημα μείωση ε, του λόγου χρέους και με αυτή τη ρήτρα που το συνδέουμε. Αν, υπε, αν κάποιος υπερβεί κατά κάποιο ποσοστό αυτό το λόγο, υπάρχουν κυρώσεις. Αλλά δεν τη συνδέουμε με το έλλειμμα. Άλλαξε δηλαδή αυτό που ενεργοποιεί το μηχανισμό, λέει ο πρόεδρος. Καρολίνα, Νάχτικα. Ευχαριστώ και τον κύριο Τίγκεσεν που ήρθε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα. Ενδιαφέρονται οι σημερινοί καιροί. Την τελευταία δεκαετία δημιουργήσαμε ένα νέο σύστημα ε, χρηματοπιστωτικό και τώρα πρέπει να το κάνουμε πιο ανθεκτικό για να έχουμε πιο ισχυρές οικονομίες. Χαιρετίζω την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Δημοσιονομικού Συμβουλίου μεν, υπάρχουν όμως πολλά που μπορούν να, ακόμη να γίνουν δε. Και έχω για κάποια ερωτήματα. Εξαιρετική καταρχάς η έκθεση, την δημοσιεύσατε τον προηγούμενο μήνα και λέτε σε αυτήν την έκθεση ότι υπήρχε προειδοποίηση σε σχέση με τις εκτιμήσεις και το τι είχε χρησιμοποιήσει ως βάση ένας φορέας. Μήπως πράγματι ήταν περιβολικές εκτιμήσεις και αυτές οφείλουν σε κάποια διαρθρωτικά προβλήματα που δεν ελήφθησαν υπόψη. Και τι γίνεται, πώς μπορεί να βελτιωθεί δηλαδή η εκτίμηση οικονομική και τι μπορεί να κάνει γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Και το δεύτερο ερώτημα για την εξάρτητη υπαρχή συμβουλών στο πλαίσιο του Συμφώνου Άπτυξης Σταθερότητας. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα σύστημα που θα έχει περισσότερα θεσμικά ε, αντίβαρα. Υπάρχει και το Συμβούλιο αυτό που μπορεί να βοηθήσει σε αυτή την κατάσταση, να βελτιώσει τα θεσμικά αντίβαρα. Μπορεί να λάβει κάποια καθήκοντα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου παραδείγματο χάρη να συντάσει τις τάσεις αναχώρα ή τις εκθέσεις αναχώρα. Αυτά είναι τα δύο. Ερωτήματα με κάποια υποερωτήματα. Uh, Ένας πρωταρχικός στόχος ε, για να λειτουργούν καλά τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια είναι να μπορούν να ελέγχουν, να παρακολουθούν τις μακροοικονομικές προβλέψεις που κάνουν οι επιμέρους κυβερνήσεις. Ορισμένα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια το κάνουν αυτό πολύ καλά, χωρίς να χρειάζονται περαιτέρω πόρους, αλλά πάλι κάνουν πιο ανεπίσημους ελέγχους των όσων κάνει η κυβέρνηση. Και γύρονται λοιπόν κάποια σημαντικά ερωτήματα τα οποία αφορούν, θεωρώ, και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν λέω ότι κάποια συγκεκριμένη εθνική κυβέρνηση μεροληπτεί στι προβλέψεις που κάνει. Στο παρελθόν έχουμε δει ότι μερικές κυβερνήσεις έχουν μεροληπτήσει. Παρ' όλα αυτά, πρόσφατα, βλέπουμε ότι οι προβλέψει ήταν θετικέ και οι προβλέψει γενικά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αξιόπιστε. Αυτό το οποίο λέμε στην έκθεση είναι μερικέ φορέ ορισμένε κυβερνήσει παρά είναι φιλόδοξε, αισιόδοξε μάλλον, όσον αφορά την οικονομική προοπτική των, δημοσίων, των δημοσίων οικονομικών του. Εμεί λοιπόν ω Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο έχουμε επικρίνει, αν θέλετε, την έλλειψη ρεαλισμού πολλέ φορέ στι προβλέψει που γίνονται. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να έχουμε πολύ υπερβολικέ απαιτήσει όσον αφορά τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια. Θα μπορούσαν όμω, αν μη τι άλλο, σε εθνικό επίπεδο να κάνουν κάποιε μελέτε και αναλύσει ε, για το πώ οι κυβερνητικέ αποφάσει επηρεάζουν ε, τι μελλοντικέ εξελίξει οικονομικέ για την κάθε χώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί απαιτεί πολύ στενέ επαφέ με την κυβέρνηση, όχι μόνο με το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και με τα Υπουργεία εκείνα που έχουν να κάνουν με διάφορε δημόσιε δαπάνε και πολλά δημοσιονομικά συμβούλια εθνικά δεν έχουν του πόρου για να κάνουν κάτι κάτι τέτοιο. Εμείς στα πλαίσια της εντολής μας προβλέπεται να διευκολύνουμε την καλύτερη δυνατή επαφή με τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια. Δεν είχαμε κι εμεί απαραίτητου πόρου για να κάνουμε κάτι τέτοιο, αλλά αυτή τη στιγμή έχει δημιουργηθεί και ένα δίκτυο εθνικών δημοσιονομικών συμβουλίων, το οποίο λειτουργεί πολύ καλά και στην έκθεσή μας θα σε δύο τέτοια εθνικά συμβούλια τα οποία κατάφεραν τελικά όντως να έχουν έναν ηγετικό ρόλο στη χώρα τους, το ένα του Ηνωμένου Βασιλείου και το άλλο της Σλοβακίας. Ιδίως στο Ηνωμένο Βασίλειο, το Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο επιβλέπει πλέον όλε τι μακροοικονομικέ προβλέψει που γίνονται από το Υπουργείο Οικονομικών. Καταλαβαίνετε ότι ο ρόλο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίω όταν προκύπτουν προβλήματα με τι οικονομικέ προβλέψει και τι οικονομικέ προοπτικέ. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν ευέλτιστε πρακτικέ που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και από τα υπόλοιπα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί βέβαια κάθε φορά που προτείνουμε ότι θα πρέπει να γίνεται με τρόπο αποκεντρωμένο ο δημοσιονομικό έλεγχο. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο συντονισμό μεταξύ των εθνικών αυτών αρχών να είναι πάρα πολύ καλό. Ξέρετε ότι μερικές φορές τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια μπορεί να είναι επικριτικά για τις οικονομικές αποφάσεις που παίρνει η κυβέρνησή τους. Μετά όμως έρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία διαπραγματεύεται με το συγκεκριμένο κράτος μέλος, λαμβάνουν συγκεκριμένε αποφάσεις από κοινού και δυστυχώς στη συζήτηση αυτή, σε επαφές αυτές δεν συμμετέχουν επίσημα τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια. Θα μπορούσαν λοιπόν να εμπλεκούν περισσότερο στην επίσημη αυτή ευρωπαϊκή διαδικασία. Νομίζω πάντως ήταν πάρα πολύ θετικό το ότι δημιουργήθηκαν τα εθνικά αυτά δημοσιονομικά συμβούλια και το ότι συμμετέχουν στην όλη διαδικασία πρόεδρο. σας. Αυτό το οποίο αναφερθήκατε, υπάρχουν δύο επιμέρους περιπτώσεις. Την πρώτη, στην πρώτη αυτή περίπτωση γίνανε κάποιες επικρίσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο και οδήγησαν σε συγκεκριμένε Αλλαγέ, ενώ στη δεύτερη περίπτωση γίνανε επικρίσεις από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, χωρίς όμως να ενσωματωθούν στις προοπτικές τη οικονομικές τη κυβέρνηση. Στη δεύτερη λοιπόν περίπτωση δεν ελήφθη υπόψη η σύσταση του Εθνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου. Από τους Πρασίνου δεν έχουμε κανέναν από την ΓΚΟΕ, από το EFDD, ο κύριο Ανεμά, από το ENF, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσω Ολλανδικά. Θα ήθελα να μιλήσουμε λοιπόν για μία ειδική περίπτωση, το Βέλγιο. Στην ετήσια έκθεση σχολιάζεται το γεγονός ότι το Βέλγιο δεν έχει εφαρμοστεί στο Βέλγιο ε, διαδικασία για την, ε, τη χρέωση του Βελγίου και ότι είναι πολύ χαλαρή ακόμα η πολιτική σε ό,τι αφορά τη χρέωση και το 3% και η σχετική διαδικασία έχει αναβληθεί για τρίτη φορά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή την χρονιά ο κύριος Γιούγκερ ανακοίνωσε ότι ξεκινώντας τη διαδικασία αυτή και πάλι λοιπόν ε, το Βέλγιο και ότι τα σχετικές ειδήσεις για το Βέλγιο είναι fake news. Πώς εκτιμάτε λοιπόν την τρέχουσα δημοσιονομική κατάσταση του Βελγίου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε την ε, στάση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και την αντίδραση του ίδιου του Βελγίου. Στο θέμα αυτό δεν είμαι η Δήμων αλλά συζητήσαμε την περίπτωση του Βελγίου. Θα πρέπει να κατανοήσουμε σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία πώς καταλήξαμε στο κάθε συμπέρασμα και στην εκάστοτε σύσταση και σε διάφορες περιπτώσεις. Ήταν δύσκολο να δούμε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις αποφασίσαμε να δείξουμε ευελεξία. Στην περίπτωση του Βελγίου υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ, ασυμφωνία μεταξύ ε, της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση του αντικτύπου φορολογικής μεταρρύθμισης για το κατά πόσο ήταν δηλαδή διαφορετικό το θέμα αυτό ή κατά πόσον υπήρχε μόνιμη αύξηση των προλογικών εσόδων. Δεν είναι λοιπόν σαφές γιατί επιλέχθηκε η εκάστοτε λύση. Ήταν ε, προσωρινή η, η λύση αυτή και δεν θα έπρεπε να έχει οδηγήσει σε χαλάρωση σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη προδιαγραφή. Αυτό λοιπόν ήταν ένα στοιχείο και γενικά πιστεύω ότι αυτό αποτελεί ένα παράδειγμα του πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει αναδόμηση, αν θέλετε, των αποφάσεων που ελήφθησαν από τις Επιπτικές Αρχές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά δεύτερον, υπήρξε και ένα άλλο παράδειγμα για μια ευρεία συμφωνία σε συστηματικό επίπεδο για την τελική αξιολόγηση. Άλλο ένα παράδειγμα του πώς προσθέτουμε ευελιξία στις πρώτες γραφές του συστήματος σε ό,τι αφορά τα δυνατότητα δηλαδή απόκλησης ε, για κάποια χρόνια. Να σας πω λοιπόν ότι δεν είμαι πεπισμένος για το ποιο είναι το σωστό αποτέλεσμα, αλλά θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να είναι πιο προσεκτική όταν ε, καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα, προκειμένου να μπορεί να αιτιολογήσει με καλύτερο τρόπο το συμπέρασμα αυτό. Αυτή είναι η τοποθέτησή μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρος και να περάσουμε στην δικασία I. Να ξεκινήσουμε με κάποιες ερωτήσεις. Θα πάρω το λόγο εγώ. Καταρχάς, για το μέλλον. Να πω ότι θεωρώ ότι η απλοποιημένη αυτή έκδοση που μας παρουσιάζεται είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ελκυστική σε ό,τι αφορά το ορόσημο των δαπανών που από ό,τι καταλαβαίνω δεν συνδέεται με το διορθωτικό έλλειμμα. Πρόκειται για μια ικανότητα που συνδέεται με τον κύκλο προσδοκιών. Ένα πρόβλημα ωστόσο εντοπίζω. Δεν είναι ίσονος σημασία όταν μας μιλάτε για το ποιο μπορεί να είναι το κληροδότημα τέτοιων μέτρων σε ό,τι αφορά το χρέος και σε, συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Λούκε αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι και μακροπρόθεσμα είναι πιο χαλαρά το μέτρο αυτό. Υπάρχει αυτό το, αυτός ο αντίκτυπος, ο αναλογικός αντίκτυπος, μιλάω και εξ ονόματο μιας κυβέρνηση ε, με ψηλή χρέωση. Άρα, αν θέλουμε να έχουμε ίσους όρους ε, ανταγωνισμού. Αν δεν επιλύσουμε τα προβλήματα που κληροδοτούνται από γενιά σε γενιά, υπάρχει πολύ άνηση εφαρμογή του συμφώνου, του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Και ιδιαίτερω αν δεν συνδεθεί αυτό με ένα σύστημα αντιμετώπιση των μακροοικονομικών ανισορροπιών, γιατί ο κίνδυνο είναι τελικά το σύστημα να είναι δυσανάλογο και να μην εφαρμόζονται στην πράξη. Για να είμαστε και Γιατί αν ήταν να ξεκινήσουμε όλοι από το μηδέν, όχι ταυτόσημοι, αλλά με ένα παρόμοιο επίπεδο χρέωσης, θα συμφωνούσα μαζί σας. Και με όσα λέτε για την δημοσιονομική ικανότητα. Σε αυτό τι έχετε να σχολιάσετε λοιπόν. Ένα δεύτερο σημείο. Μία παρατήρηση, μάλλον. Η αξιολόγησή σας για την διάταξη ευελιξία στο 2017 που διέφερε από αυτή το 2016. Έχουμε τρία ουσιαστικά επίπεδα. Έχουμε την επικοινωνία σε θέματα επενδύσεων, έχουμε τις διατάξεις για τα αναπάντεχα πρέαστικά και ε, έχουμε και κάτι το οποίο είναι εκτός ε, της ευελιξίας, αλλά όπου πάλι εφαρμόζονται οι κανόνες. αξιολογήσατε το ποια θα ήταν η δημοσιονομική κατάσταση των κρατών μελών χωρίς τη ρήτρα αυτή. Τι θα είχε γίνει δηλαδή σε περίπτωση που δεν είχε χορηγηθεί αυτή η ευελιξία σε συνολικό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών. Και τρίτη παρατηρήση. Είμαστε σε ένα δύσκολο σημείο σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία του δημοσιονομικού μας προγράμματος ενώπιον ουσιαστικά μιας πρόκλησης, μιας μεγάλης πρόκλησης. Άρα, Νομίζω ότι υπάρχει κάποια αξία στο να μπορούμε να επιτύξουμε ότι μπορεί να εφαρμοστούν οι κανόνες με κάποια ευελιξία. Γιατί αυτό καταδεικνύει ότι δεν μπορούμε απλά να απορρίψουμε εφάπαξ τους ε, κανόνες. σε ό,τι αφορά την ε, τήρηση των κανόνων με κάποιες διαφορετικές ε, αποκλήσεις, γιατί εδώ μιλάμε για χρόνια και ποσοστά τέτοια. Δεδομένης λοιπόν της κατάστασης, μήπως αναθεωρείται την κριτική στάση που τηρήσατε σε ό,τι αφορά το 2016 και 2017 και την ευελιξία. Έχετε δίκιο ως προς το ότι το θέμα της κληρονομιάς ίσως ε, το χρέος δηλαδή δεν το έχουμε μέχρι τώρα ίσως ε, εκτιμήσει επαρκώς. Ε, υπήρχαν χώρες με 130% χρέος και το 60% είναι κάτι πολύ μακρινό, μακροπρόθεσμο. Οπότε άλλοι κανόνες, άλλες συνδείξεις ε, χρειάζονται ίσως. Και σίγουρα υπάρχουν ε, επικίνδυνες επιπτώσεις ε, της μουσουλμικής πολιτικής από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Τώρα κοινοί δημοσιονομικοί κανόνες δεν είναι κάτι που το σκεφτόμαστε. Ίσως ήταν οι επιπτώσεις περιορισμένες, αλλά αν τα επίπεδα χρέους είναι μεγάλα, είναι πολύ σημαντικές επιπτώσεις αυτές. Πρέπει να υπάρχουν κανόνες μείωσης του χρέους σύν το χρόνο. Αν διαβάσετε την πρότασή μας, είναι μια ήπια πρόταση νομίζω. Αυτό με τον των κανόνων ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό. Έχετε δίκιο. Απλά υπάρχει αυτός ο κύκλος των κανόνων. Κάποιοι κανόνες το 11-13 ήταν πολύ αυστηροί. Παντού σχεδόν τότε είχαμε στην Ευρωζώνη ύφεση. Τότε χρειαζόταν ευελιξία, αλλά υπήρχε μεγάλη νευρικότητα. Και ήταν πολύ επικίνδυνη κατάσταση για να εφαρμοστεί τότε ευελιξία. Η ευελιξία εφαρμόζεται όμως όλο και περισσότερο, από το 15 και μετά τουλάχιστον. Και όλο και περισσότερο όταν χρειάζεται και πολύ λιγότερο κατά την άποψή μου αυτή η ευελιξία. Έχετε λοιπόν δίκιο ότι είναι με εξαίρεση κατά κάποιο τρόπο. Και το αποτέλεσμα ήταν χαμηλότερα ποσοστά ανάπτυξη και στην Ευρωζώνη. Σίγουρα χρειαζόταν αυτή εκτακτή δόση ευελιξίας τότε βέβαια. Ε, Δείχνει δεκτές και παρεκκλήσεις από τους κανόνες. Έχουμε ένα πίνακα στο κεφάλαιο 5 και εκεί συνοψίζουν. Και το τι έγινε στην Ιταλία. 2 με 2,5% το ΕΠ το 15, 16, 17. Μπορεί λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση να ήταν σωστά το μέτρο, αλλά σε κάποιε άλλε χώρε ίσω να μην ήταν τόσο. Ασκήσαμε κάποιε κριτικέ, κάποιε επικρίσει. γιατί λέμε και πιστεύουμε ότι η ευελιξία στου κανόνε είναι μια πρακτική που εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση. Την εκάστοτε δεν εφαρμόζεται σταθερά ή προκυκλικά, όπω έγινε το 17 κατά την απόψή μα και ίσω και το 18 χωρίς να θέλω να προτρέξω στο τι θα περιλαμβάνει η έκθεσή μας για του χρόνου. Ε, έχετε δίκιο ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση σε αυτή την όλη λογική των κανόνων, αλλά νομίζω ότι η πολύ ανοιχτή ερμηνεία ή πολύ αυστηρή ανάλογα με την περίοδο δημιούργησε προβλήματα. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλο το λόγο. Ντανούτα, θέλεις το λόγο. Ε, άντε, ένα λεπτό. Ναι, γιατί δεν έχουμε μιλήσει για τα εθνικά επίπεδα, αλλά στην έκθεση, και στην έκθεση σας δεν λέτε και τίποτα. Τι μπορεί να γίνει σε εθνικό επίπεδο για βελτίωση της κατάστασης ή για να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία σε ό,τι αφορά αυτό το δημοσιονομικό πλαίσιο τώρα έχουν περισσότερο χρόνο για να εντάξουν τη στάση του στην Εθνικά Κοινοβουλή σε σχέση με το παρελθόν. Θεωρείται όμω ότι απαιτούνται και άλλε αλλαγέ για να βελτιωθεί ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί αυτό το δημοσιομικό πλαίσιο σε εθνικό επίπεδο. Μπορούν να γίνουν περισσότερα ή πρέπει όλα να βελτιωθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κοιτάξτε, είναι δύσκολο να απαντήσω την ερώτηση αυτή γιατί σαφώς μπορεί να γίνουν περισσότερα πράγματα σε εθνικό επίπεδο, αλλά είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί. Ορισμένοι δυσκολεύονται να καταλάβουν για ποιο λόγο έχουμε συγκεκριμένους δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι δεν θα πρέπει να ειδωθούν ως κλωβός, ως ζουρλομανδίας που εγκλωβίζει τα κράτη-μέλη, αλλά ως κάτι υποφελία τους πάντες. Είναι πολύ σημαντικό όμως και τα εθνικά δημοσιονομικά συμβούλια να μπορούν να κάνουν συστάσεις και αν ήταν πιο έντονη η συμμετοχή τους, τότε πραγματικά θα μπορούσαμε να κάνουμε και προβλέψεις λίγο πιο μακροπρόθεσμες, οι οποίες θα έρχονταν από το εθνικό επίπεδο και θα πήγαιναν προς το ευρωπαϊκό επίπεδο. Προφανώς εγώ θα ήθελα και μεγαλύτερη συμμετοχή και από τα εθνικά κοινοβούλια, αλλά έχω την εντύπωση ότι τα προσχέδια προπολογισμού και όλα αυτά τα έγγραφα τα οποία υποβάλλονται στο πλαίσιο του προγράμματος σύγκλησης τελικά δεν συζητώνται ή δεν συζητώνται επαρκώς στο πλαίσιο των εθνικών κοινοβουλίων. Νομίζω λοιπόν ότι θα έπρεπε και τα όργανα αυτά να συμμετέχουν περισσότερο και είναι κρίμα που δεν συμμετέχουν. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πολύ χρήσιμη και επικοδομητική και πλούσια θα έλεγα αυτή η ανταλλαγή απόψεων και προφανώς και το κοινοβούλιο μας αυτό και το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα συνεχίσει το σημαντικότατο αυτό διάλογο που έχουμε ξεκινήσει με το Ευρωπαϊκό Δημοσιονομικό Συμβούλιο προκειμένου να βελτιώσουμε τους δημοσιονομικούς μας κανόνες και να καταφέρουμε να βελτιώσουμε γενικότερα τη διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Σας ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την έκθεσή σας, για την παρουσία σας εδώ και προσβλέπουμε στην επόμενη ανταλλαγή απόψεων. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Next item. Περνάμε στο επόμενο σημείο λοιπόν της ημερήσιας διάταξης. Εδώ προβλέπεται η συζήτηση της γνωμοδότησης τη κυρία Ιβάνα Μαλέτιτς όσον αφορά την πορεία της συζήτησης για το μέλλον της Ευρώπης. Προβλέπεται συγκεκριμένη εξέταση των τροπολογιών. Ιβάνα, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους σκιώδεις εισηγητές, καθώς επίσης και όλους τους συναδέλφους που κατέθεσαν τροπολογίες δεν ήταν ε, σε καμία περίπτωση εύκολο να καταλήξω σε συμβαστικέ προτάσεις γιατί για συγκεκριμένα σημεία αποκλείουν πολλοί απόψεις μας. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι στην επόμενη συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τις συμβαστικές τροπολογίες. Κάποια παραδείγματα τώρα. Κάτι το οποίο είναι πολύ θετικό καταρχάς είναι ότι έχουμε συμφωνήσει για τα βασικά ορόσημα, θέλετε, της γνωμοδότησης αυτής, τα οποία θα πρέπει να εμπεριέχονται σε αυτή τη γνωμοδότηση σε κάθε περίπτωση. Λέμε ότι θα πρέπει να καλύψουμε όλα τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής και όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία ξεφεύγουν, αν θέλετε, λίγο από τις δικές μας αρμοδιότητες, θα πρέπει να βρούμε μια κάποια θέση στις συμβαστικές τροπολογίες αλλά δεν είναι απαραίτητο να καλύψουμε τα στοιχεία αυτά πλήρως. Δεν αποτελεί αυτό απόλυτη προτεραιότητα και φαντάζομαι ότι θα δείξουν προ προς αυτό κατανόηση οι συνάδελφοι. Όσον αφορά την Τραπεζική Ένωση, υπάρχει εδώ πέρα μια διαφορετική προσέγγιση από κάποιους συναδέλφους. Θα θέλανε μια πιο σταδιακή ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης σε σχέση με την άλλη άποψη που προβλέπει μια ταχεία ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Επίσης υπάρχουν διαφορές στις απόψεις μας όσον αφορά το SBPS και τους σχετικούς κανόνες. Θα δούμε στην επόμενη συνεδρίαση πώς θα καταφέρουμε να απευθυνθούμε στο ζήτημα αυτό. Έπειτα, Ένωση Κεφαλαγορών. Εδώ θέλουμε να εμπλέξουμε λίγο περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να λέμε πόσο σημαντική είναι τελικά η Μελλοντική Ένωση Κεφαλαγορών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, γιατί θα έχουν κατά αυτόν τον τρόπο μια επιπλέον πηγή χρηματοδότησης οι εταιρείε αυτές. Όσον αφορά τώρα τη δικασία τη εμβάθυνση και τη ολοκλήρωση τη οικονομική και Νομισματική Ένωση, ω προ αυτό έχει γίνει μια πρόταση για το ότι θα πρέπει να έχουμε μια δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωζώνης, ότι αυτό είναι θετικό και ότι θα πρέπει να έχουμε και νέους δημοσιονομικούς κανόνες όσον αφορά τη σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, καθώς επίσης και ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανεργίας σε επίπεδο Ευρωζώνης. Αυτό δεν προτείνεται ακόμα επίσημα, επίσημα στο κείμενο και έχουν γίνει και άλλες σχετικές προτάσεις που έχουν να κάνουν με την ενίσχυση των ε, ε, επενδύσεων και άλλα ε, χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία θα μπορούσαν και αυτά να συμβάλλουν στην δημοσιονομική ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωζώνης μάλλον. Ελπίζω να καταλήξουμε και εδώ σε καλούς εμβιβασμούς. Τέλος, είπαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε και το πρόγραμμα στήριξης των δραστηριοτικών μεταρρυθμίσεων. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που είναι υπέρ του προγράμματος αυτού, άλλοι πάλι που δεν θέλουν να υποστηρίξουν το πρόγραμμα αυτό, αλλά που θα θέλανε περισσότερο να υποστηρίξουν την ε, ε, λειτουργία σταθεροποίησης ε, των ευρωπαϊκών οικονομιών μέσω των επενδύσεων. Επίσης, πρέπει να αποφασίσουμε και για τη συγκεκριμένη πρόταση που θα κάνουμε για το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, αν θα πρέπει να αναθεωρηθεί ή αν θα πρέπει να εξακολουθήσουν να ισχύουν οι υφιστάμενε ρήτρε ευελιξία που περιέχονται στο σύμφωνο αυτό, οι οποίε όμω, αναγνωρίζουν περισσότεροι συνάδελφοι, δεν εφαρμόζονται σωστά στην πράξη. Μεγαλύτερη διαφάνεια επίση και καλύτερο σύστημα επικοινωνία και ενημέρωση προ Ευρωπαίου πολίτε. Ω προ αυτό συμφωνούν οι περισσότεροι συνάδελφοι. Σα ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Περβάνς Μπερές. Ευχαριστώ. Η πρώτη φορά ε, που είμαι σκιώδης για αυτή τη βδομάδα ε, αντί του σκιώδους, ε, να δω πόσους άλλους αντικαταστήσω αυτή τη βδομάδα, αυτή τη σημαντική αντικαταστήσω τον Κώστα Μαυρίδη που δεν μπορούσε να είναι εδώ. Θα ήθελα να κάνουμε καταρχάς μια οριζόντια παρατήρηση ό,τι αφορά την έκθεση της συναδέλφου Έχουμε και την έκθεση του συναδέλφου μας ε, Ραμόν Χαρέιτη που έχει να κάνει το μέλλον της Ευρώπης, ε, πολύ σημαντική. Εμείς ε, γνωμοδοτούμε για αυτήν την έκθεση και δεν έχω κάποιο πρόβλημα με αυτό, αλλά βλέπω ένα κίνδυνο στη ζήτηση που μόλις ξεκίνησε. Με εκθέσεις δηλαδή πρωτοβουλίας που γνωμοδοτεί η Επιτροπή μας, να έχουμε τελικά αξιολόγηση πολύ συγκεκριμένων προτάσεων που είναι επιτάπητος. και που μπορεί να έχουμε δύο διαφορετικέ απόψει για ένα θέμα που όμω δεν έχει κλείσει. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να κλείσει το ε, θέμα αυτό όταν ψηφίσουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Εμείς έχουμε τη ομάδα από την Επιτροπή μας, ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και αυτό που λέω αφορά αρκετές προτάσεις. Να σας πω μερικές από αυτές. Το InvestEU. Η σταθεροποιητή λειτουργία, προστασία των επενδύσεων, το πρόγραμμα υποστήριξη κτλ. Και άλλα. Σας λέω αυτά τα τρία παρόδο. Και έχω έψει ανησυχίε. Μήπως τελικά καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που να είναι πιο οριστικός κατά κάποιο τρόπο όπως θα θέλαμε. Εγώ θα έλεγα να έχουμε ώστε να το μια πιο γενική προσέγγιση που μπορούν να την υποστήριξουν περισσότεροι. τι ήθελε τώρα συγκεκριμένα να πει ο Κώστας Μαυρίδης. Το θέμα της ολοκλήρωσης της Τραπεζικής Ένωσης σίγουρα είναι σημαντικό. Πρέπει να αναφέρεται η πλήρης ε, ε, Τραπεζική Ένωση και το έντις. Εδώ και καιρό το θέλουμε αυτό. Δεύτερο. στο πλαίσιο τη συζήτηση για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Εξαμενού. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη νέα διάσταση, αλλά δεν έχουμε πολλά στοιχεία τη στην πρόταση αυτή. Όπω παραδείγματο χάρη, βιώσιμη ανάπτυξη. Και πώ ο μετασχηματισμό που γίνεται σε οικονομικό, κοινωνικό, περιβαλλοντικό επίπεδο θα πρέπει να ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο. Τρίτον, Έχουμε τον Ευρωπαϊκό Πυλόν Ανθρωπίνων, ε, Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Πάνω σε αυτόν πρέπει να εστιάσουμε. Μπορεί κάποιοι να πούνε ότι δεν είναι ε, στη δική μας, ε, της δικής μας αρμοδιότητας. Η ΕΜΠΛ δυστυχώς όμως δεν γνωμοδοτεί από ό,τι είδα. Εμείς ως Επιτροπή Οικονομικών Αποθέσεων πάντοτε λέμε ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η κοινωνική διάσταση της ΩΝΕ. Άρα δεν θα πρέπει να παραγνωρίσουμε αυτή τη διάσταση εντελώς. Σε ό,τι αφορά τώρα την καταπολέμηση των αποκλήσεων, ναι, είναι σημαντικό, πρέπει να το δούμε. Αυτό πιστεύει και ο σκιώδης μας, ο Κώστας Μαυρίδης. Τα νέα εργαλεία τώρα. Νομίζω τα στηρίζει επί της αρχής, αλλά αναφέρω ξανά την παρατήρηση που έκανα στην αρχή ότι θα πρέπει να προδικάσουμε και την έκφραση των διαπραγματεύσεων, γιατί υπάρχουν πολλά θέματα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Και τέλος, ό,τι αφορά το Ταμείο Συνοχής θα ήθελε να επενθυμίσει τι ψηφίσαμε ήδη στην Επιτροπή μας. Δηλαδή τη διασύνδεση με την μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Δεν είναι κάτι που στηρίζουμε. Η έκθεση αυτή θεωρεί πάντως ότι είναι πολύ σημαντική. Ένα χρόνο πριν τις ευρωεκλογέ. Και φυσικά είναι και πρόθυμος να συνεισφέρει στην επίταξη καλού συμβιβασμού. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος. Δεν βλέπω άλλους κοιόδης. Ποιος άλλος θα θέλει τον λόγο. So after... Μετά τους όδης λοιπόν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ραμόν Χάουρικ. Παρεμβαίνω στο πλαίσιο τη διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑ γιατί συνεργάζομαι με την κυρία Μάλετιτ στο πλαίσιο τη έκθεση αυτή και θέλω να την ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα για τη συνεισφορά στην έκθεση αυτή, όπω έλεγε και η Περβάν Μπερέσε στην ΑΦΚΟ, που είναι η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή, εκπονούμε μια έκθεση που ίσως κάπως φιλόδοξα την ε, ονοματίσαμε μέλλον της Ευρώπης. Ε, το μέλλον της Ευρώπης σίγουρα δεν το έχουμε γράψει ακόμη, ε, είναι σε εξέλιξη ο προβληματισμός ο σχετικός. Αλλά στη Συνταγματική Επιτροπή θέλουμε να επικαιροποιήσουμε όλα τα έγγραφα και όλες τις συζητήσεις που γίνονται τα τελευταία χρόνια εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινούβολο και όχι μόνο. Γενικώ συζητείται το θέμα αυτό, το μέλλον της Ευρώπης. Σίγουρα υπάρχουν τα ε, γνωστά ότι δεν είναι πλήρης η λειτουργία, υπάρχουν ατέλειες, μπορεί να βελτιωθεί, αλλά υπάρχει και ένα ε, κεφάλαιο που έχει να κάνει με το οικονομικό σκέλος. Η Σταγματική Επιτροπή τι θέλει. Η ΕΚΟΝ, η Επιτροπή σας δηλαδή αυτή, να πει πραγματικά ποια είναι τα βασικά στοιχεία, οι βασικές γραμμές για την ε, οικονομική πολιτική. Είναι η Επιτροπή σα αυτή που είναι στην καλύτερη να τη θέση για να το πράξει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα με την κυρία Μάλιτιτ και στις ε, συζητήσεις που θα έχουμε με τους Κιώδης να δούμε με ποιο τρόπο η ΕΚΟΝ θα καταθέσει προτάσεις που θα βρουν ε, πλήρη υποστήριξη στην Επιτροπή έχουμε και το κανόνα 54 που θεσπίζει τη συνεργασία ΕΚΟΝ για το θέμα αυτό και εμείς αυτό που θέλουμε είναι η έκθεση της ΕΚΟΝ, η γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ να ενσωματωθεί πλήρως στην έκθεση της Επιτροπής Ταγματικών Υποθέσεων. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό λέω σωστά τα είπε και η κυρία Μπερές. Η πρόθεσή μας δεν είναι στην έκθεση να απαριθμίσουμε εξαντλητικά όλες τις λύσεις για το κανονικό μέλλον της Ένωσης. Όμως αυτό που λογικά θέλουμε είναι να μας ε, δώσει κάποιες γενικές, κάποιες αδρές γραμμές για τα μείζωνα θέματα. Από οικονομικής, χρηματοπιστωτικής πλευράς, ε, τα θέματα που εκκρεμούν ακόμη, διακυβέρνηση τη ΟΝΕ, Τραπεζική Ένωση, Δημοσιονομική Πολιτική, Δημοσιονομικό Πολιετές πλαίσιο, οι δίποροι, προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωσης, για όλα αυτά τα θέματα και πάλι δεν έχουμε την πρόθεση να ξεκινήσουμε νέες συζητήσεις ε, με πρωτοβουλία της ΕΚΟ. Όχι, απλά υπάρχουν έγγραφα τα οποία έχετε εκπονήσει και πρέπει να ληφθούν υπόψη. Αυτός είναι ο στόχος και δράτω με τις ευκαιρίες που μας προσφέρει αυτή η συζήτηση για να πω ότι η Συνταγματική Επιτροπή αυτό που θέλει είναι να ενσωματώσει στο σύνολό της τη γνωμοδότηση της ΕΚΟΝ. Και σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι προτίθεμαι και διμέρως να συνεργαστώ με την κυρία Μάλετιτς, την οποία ευχαριστώ για τη συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Άλλη. Um, so please, uh, Η παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω ότι είναι πολύ θετικό το γεγονό ότι είναι καλή η συνεργασία με την Επιτροπή Στεγματικών Υποθέσεων και με την εισηγήτρια, τον εισηγητή, τη ΑΚΟ. Ελπίζω στο τελική ανάλυση να μπορέσουμε να συνδυάσουμε την άποψή μα και τι προτάσει που έχουν ήδη συμπεριληφθεί στην έκθεση τη Επιτροπή Στεγματικών Υποθέσεων και αυτό γιατί υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία έχουν να κάνουν με ζητήματα αρμοδιότητας της οίκων. Νομίζω ότι θα καταφέρουμε να συμφωνήσουμε επ' αυτόν. Συμφωνώ επίσης ότι ενδεχομένω καλύτερο θα ήταν να μην προσπαθήσουμε στη γνωμοδότηση αυτή να ολοκληρώσουμε κάτι το οποίο καλύτερα να συζητηθεί σε διάφορους φακέλους, σε διάφορα θέματα, αλλά αυτό δεν είναι πάντα εύκολο όταν μιλάμε για την ε, Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση και την ανάγκη εμπάθησης αυτής και για την σύγκληση των κρατών μέλων στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναφέρουμε ένα πρόγραμμα υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων σε ό,τι αφορά και τη δυνατότητα υποστήριξη ε, τη σύγκληση στι ε, χώρε που δεν είναι στην Ευρωζώνη. Ελπίζω λοιπόν στην τελική ανάλυση να καταφέρουμε να το ξεκαθαρίσουμε αυτό στην ε, γνωμοδότηση Και επίσης αυτό που αναφέρετε και εσείς κυρία Μπρές, αναφορικά με την άποψη του κυρίου Μαυρίτη για τα ταμεία συνοχής, ότι θα πρέπει να μπει στην ε, γνωμοδότηση ότι δεν χρειάζεται αυτή η σύνδεση με τη μακροοικονομική αιρεσιμότητα. Νομίζω ότι καλύτερα θα ήταν να το δούμε αυτό στο φάκελο στο θέμα CPR. Γιατί Δεν έχουμε το σύνολο του κανονισμού εδώ. Και αναφέραμε και τα θέματα βιώσιμη ανάπτυξη, κλιματική αλλαγή, κοινωνικών δικαιωμάτων. Ελπίζω να μας ικανοποιούν όλα αυτά. Και θα δούμε πώς θα εταιρεθεί αυτή η πιο γενική προσέγγιση, όπου αυτό ασφαλώς είναι δυνατόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Ζητήσατε το λόγο. Εξέταση των τροπολογιών έλαβε χώρα σήμερα. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα στις 19 Νοεμβρίου. Σε ό,τι αφορά αυτά που είπε η κυρία Ατούντο, εν ώψη της Προεδρίας αναμένουμε ότι η Επιτροπή Σταγματικών Υποθέσεων θα εξετάσει το θεσμικό πλαίσιο για τη Σύμβουλη της εικόν. Άρα υπολογίζουμε σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα οι ψηφοφορίε. Να κάνουμε λοιπόν ένα διάλειμμα 10 λεπτών. Ευχαριστώ. So, dear colleagues, uh, please. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε σας παρακαλώ πολύ. Θα κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίστε, ψηφίζουμε δοκιμαστικά. Καταφθάνουν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι. Okay. 39. Okay. We close. Πολύ ωραία πέρας της ε, δοκιμαστικής αυτής προφορίας. Διαδικαστικό από την Περβόνς παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε μια έκθεση που έχει να κάνει με τις διασυνοριακές πληρωμές και είδαμε από την αρχή του απογεύματος μπροστά στην αίθουσα αυτή λομπίστες οι οποίοι είναι υπέρ της δικής τους βέβαια θέσης και δίνανε και κάποια έγγραφα ντεπλιάν, φυλάδια κτλ. Στους βουλευτές που μπαίνανε στην αίθουσα αυτή προσπαθώντας να τους δώσουν κάποια κατεύθυνση για τον τρόπο που θα πρέπει να ψηφίσουν. Νομίζω ότι αυτό αντιτίθεται εντελώς στην εντολή που έχουμε ως ευρωβουλευτές Μπορούν να κυκλοφορούν οι άνθρωποι αυτοί βέβαια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι ποτέ δυνατόν να αποδεχθούμε ότι τη στιγμή που ετοιμαζόμαστε να ψηφίσουμε, να έχουμε μέλη ομάδων πίεση οι οποίοι μα λένε τελευταία στιγμή πώ θα πρέπει να ψηφίσουμε. Αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε και συμφωνώ μαζί σας ότι δεν είναι σωστό κάτι τέτοιο. Θα ζητήσω λοιπόν από τη Γραμματεία να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει ενδεχομένω του λομπίστε που κάνουν κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Οι κανόνε μα είναι σαφεί, θα πρέπει να τηρούνται και στου κανόνε αυτού προφανώ δεν περιλαμβάνεται η διαφήμιση πρόθεση συγκεκριμένων πολιτικών θέσεων έξω από τη δική μας την αίθουσα ενώ ετοιμαζόμαστε για ψηφοφορία. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με την ψηφοφορία και την έκθεση του Ashley Fox όσον αφορά τους Ευρωπαίους Πάροχους Υπηρεσιών Πλήθο Χρηματοδότησης για Επιχειρήσεις 137 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 184 ως την 186 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. Τροπολογίες 188 και 189 από κοινού υπέρ, κατά. ηλεκτρονική επαλήθευση, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρασε απορρίπτονται 27 έως μάλλον η τροπολογία 29 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 190 και 198 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται συμβαστική τροπολογία α υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 196 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 38 υπέρ κατά 31 διορθώνω πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Β πρώτο τμήμα υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ παρακαλώ κατά Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 45. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 219 και περνάμε στη συμβαστική I, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 28 υπέρ, διορθώνει ο Πρόεδρος, Πρέπει να ψηφίσουμε και κάποιες άλλες τροπολογίες. Τροπολογία 70 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 262 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συνεχίζουμε. 135 και 131 μαζί υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτονται. 187 υπέρ παρακαλώ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. 220 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Να ψηφιστεί μόνο αν η συμβαστική I έχει εγκριθεί, λέει ο Πρόεδρος. Συμβαστική J. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Άρα ψηφίσουμε την 71 και τη 265 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 266 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 264 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 267 υπέρ κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική C υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 224. Δεν την ψηφίζουμε, λέει ο πρόεδρος, μάλιστα. Περνάμε στην τροπολογία 49. Υπέρ, παρακαλώ. κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Ι e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική, μάλλον τροπολογία 235 υπέρ. Το είπα. Τροπολογία 235. Ο πρόεδρος είπε κατά λάθο συμβαστική 235. Ψηφίσουμε την τροπολογία 235 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 235. Άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβαστική G υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 238 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 238, άρτη ψηφοφορία. Πέρασε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 239 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τη συμβαστική H, άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε έτσι στην τροπολογία συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 226 πέρα. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση τροπολογία 226. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 282. Αυτή καταπίπτει μάλλον. Α πάμε συμβαστική N υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική O υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P. Πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Μάλλον ηλεκτρονική επαλήθευση για το πρώτο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας π. Άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της συμβαστικής π. Υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 316 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική R πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλλον όχι. 109 υπέρ κατά αποχές. Το έλκυνε κατά τις 109. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 109 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 23 υπέρ 20 κατά. 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή. Υπέρ Κατά. Το ΕΛΚ για την προφορική τροπολογία στην ΠΕΡΑ. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 111 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η 111. Συμβαστική ΑΑ υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται. 115 τώρα, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική AB, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 με προφορική τροπολογία από τον εισηγητή, με δύο προφορικές τροπολογίες μάλιστα, όχι μία μόνο. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την 132 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται 24 υπέρ 20 κατά. Ψηφίσουμε τώρα από κοινού την 133 και την 134 υπέρ κατά αποχές το υπέρικατα. υπέρ ή κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση για τις 133 και 134 άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτονται. Συμβαστική S υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 333 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές εγκρίνεται 334 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία T υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική U υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 145 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 147 υπέρ ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 147 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 25 κατά 19 υπέρ, 148 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Β, υπέρ, κατά αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 156, υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 157 υπέρ, κατά αποχές, απορρίπτεται. 158 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 159 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία Z υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρα πρέπει να ψηφίσουμε όλες τις υπόλοιπες 151 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 160 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 150 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 163 υπέρ κατά ηλεκτρονική επαλήθευση για τροπολογία 163 άρτη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Η οκτώ είναι συμβατή. Υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία W. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία X. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 11. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 173 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Y υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. προπολογή 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 26 και 180 και 181 και οι τρεις μαζί. Όχι, 26 και 180 μαζί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται 181 υπέρ. Μάλλον καταπίπτει 181, 182 έχει αποσυρθεί. Περνάμε στην 27 και την 183 μαζί. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με ονομαστική κλίση άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίνεται 38 υπέρ, 5 κατά, καμία αποχή. Ψηφίζουμε για την απόφαση να ξεκινήσουμε διοργανικές διαπραγματεύσεις, μονομαστική κλίση, άρτη ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. 38 υπέρ, 4 κατά και 2 αποχές. Έχουμε λοιπόν την ειδική πλειοψηφία που απαιτείται. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. We move to the next. Crowdfunding 2. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα για το crowdfunding. 2. Καρολίνη Νάχτεχάλα. Συμβαστική C αγορέ χρηματοπιστωτικών δικο μέσων. Υπέρ κατά λοιπόν αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2. B. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική α. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία για την αιτιολογική σκέψη 2. Υπέρ κατά Απόχε εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία στο αιτιολογική σκέψη 3. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ψηφίζουμε στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε με μονοδική κλίση. Παρακαλώ ψηφίζουμε. Πέρασε. 41 υπέρ, 2 κατά, Εγκρίνεται. Και τώρα για να ξεκινήσουν παρακαλώ η ψηφοφορία για την ε, κίνηση των διεθνικών ε, διαπραγματεύσεων ψηφίζουμε. Πέρας. 40 υπέρ, 3 κατά, 0 απόχεια. Συγχαρητήρια στην συγκεκριά. επόμενη έκθεση για τη βιώσιμη χρηματοδότηση. Πολ Τάγκ. Γνωστοποίηση σχετικά με τι αηφόρε επενδύσει. 47 τροπολογία υπέρ. Κατά. Το ΕΛΚ είναι υπέρ, παρακαλώ. Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική Α υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 109 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές Έλεγχος παρακαλώ για την 19. Πέρας. Απορρίπτεται 21 η ψήφη κατά 18 υπέρ. Συμβαστική C υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε δεύτερο τμήμα υπέρ. Έλεγχος παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτεται οι ε, 16 ψήφοι υπέρ 23 κατά. ψηφίσουμε λοιπόν την 181 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται. 180 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική G. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΙΤΑ H υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιώτα αι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 228 υπέρ κατά. Έλεγχος. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. Απορρίπτεται 22 ψήφοι κατά 21 υπέρ. 229 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 230 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 231 και 233 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 232 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 235 και 236 υπέρ κατά έλεγχος παρακαλώ ηλεκτρονική επαλήθευση Πέρας. Απορρίπτεται. 22 κατά 20 υπέρ. Τροπολογία 237. 237 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 231 με προφορική τροπολογία της κυρίας Πιτικάινεν. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική F υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική M μη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική N νη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ομικρόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική P ε, ε, ρο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική Q υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική R υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική S υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 7 με προφορική τροπολογία της εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 79 υπέρ κατά. Έλεγχος, παρακαλώ. Ελέγχουμε την 78. Πέρας. Απορρίπτεται. Η συμβαστική τάφη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική γιου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποστροποποιήθηκε, Η ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρας. 41 ψηφί περ 2 κατά 0 αποχές. Τώρα να ψηφίσουμε για την απόφαση έναρξης διαπραγματεύσεων στα πλαίσια τριμερούς διαλόγου. Με ονομαστική κλίση ψηφίζουμε. Πέρασε. 39 ψήφοι, υπέρ, 2 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Και τώρα να περάσουμε στην έκθεση της κυρίας Εύας Μάιντελ για τις διασυνοριακές ε, συναλλαγές. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική μείον α καινούριο φρούτο αυτό. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική α, κανονική αυτή τη φορά. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική B, Β, υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική D υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική ε e, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά απορρίπτεται. Αποχές απορρίπτεται, συγγνώμη. Συμβαστική G. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική H υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική I υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική J υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική K υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική L υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική O, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα ψηφίζουμε την ούτως τροποποιηθή σαν πρόταση της Κομισιόν ονομαστικά. Άρχεται η ψηφοφορία. is closed. Πέραση ψηφοφορίας. 37 υπέρ, 3 κατά και 3 αποχές. Ονομαστικά την απόφαση για έναρξη τριμερούς διαλόγου. Ονομαστικά επαναλαμβάνω. Πέρας ψηφοφορίας. 38 υπέρ και 5 κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτριά μας. Ολοκληρώσαμε λοιπόν επόμενη συνεδρίαση Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα. Πέρα της συνεδρίασης.